Ξεκινώντας θα ήθελα να κάνω ορισμένες ε, παρατηρήσεις σχετικά με τις δηλε... Ε, γραπτές δηλώσεις που έχουν παρουσιάσει οι συνάδελφοι Μακταρα Ραμπέλα Ρετζίνα Μπάστος, Πασκάλ Κάνφιν, Μαρή Κριστίν Βερσιά, Ρενάτ Βέμπερ ως προς τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Καθεστώτος ε, Καταστατικού για την αλληλασφαλιστική εταιρεία, τον συνεταιρισμό και το Ίδρυμα που έχει συλλέξει τις υπογραφές της πλειονότητα των μελών που αποτελούν το Κοινοβούλιο και άνω και ως εκ τούτου θα κατατεθεί βάσει του άρθρου 123 του κανονισμού μας στις αρμόδιες αρχές και θα δημοσιευθεί στα σχετικό έντυπο. Η γραπτή δήλωση των ε, κυρίων Φιώνα